Can we start the meeting? Thank you. Thank... Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα καλύπτονται όλες οι γλώσσες. Ε, πλην της Ιρλανδικής γλώσσας βεβαίως από ό,τι βλέπω στις μου δεν μπορείτε να μιλήσετε, λυπάμαι. Σήμερα θα εκλέξουμε πρόεδρο για την Επιτροπή Απασχόλησης. κάποια μέλη συμμετέχουν ως αναπληρωματικά ε, στην ε, συντριπτική αυτή επιτροπή. Ο κ. Λαουτού από τους Χριστιανούς Δημοκράτες ε, αντικαθιστά την κυρία Ντόμπροφ κυρία Λάνα Καλπεσμούνιος, τον Νίλς Σούκοσαν. Επίσης, άλλος συνάδελφος καλύπτει την κυρία Γαλιάνη, εκτός και αν είναι εδώ ήδη. Ευχαριστώ. Μαρή Πιέρ Βεντρέν. Αντικαθιστά ο Γιάνν Μπόντρι. Γιώργη Κάνας αντικαθιστά την κυρία Ράτκα Μάξοβα. Ανδρέα Κάροπο αντικαθιστά την κυρία Στεφάνα Σαμπέλη. Η κυρία Τζούλη Λασαντέι την Σφραν Κέμετ. Και σκύρεντα από το ΕΛΚ αντικαθιστά το κύριο Τόμακ. Και στη συνέχεια θα αποχωρήσει ο κύριος Βίλεμσον και θα την αντικαταστήσει ο κύριος Κουσμόα από την ΚΟΕ. Ωραία, κηρύσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης να σας πενθυμίσω και πάλι ότι σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι να συγκροτηθεί το Προεδρείο σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων, σύμφωνα με τον κανόνα 2.1.3. Πρώτα θα εκλέξουμε Πρόεδρο και μετά αντιπρόεδρο. Λοιπόν, απαρτία έχουμε. Και τώρα έρθει η ώρα να ακούσουμε τις υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Βίκτορ. Ευχαριστώ. Είμαι εδώ ως συμπρόεδρος της ομάδας του ECR για να προτείνω την υποψηφιότητα ε, του συναδέλφου, της συναδέλφου Σίσλο. Το κάνω για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος ε, είναι λόγω του πλήρους ε, σεβασμού της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, γιατί εδώ Εκπροσωπώ μια πολιτική ομάδα που αποτελείται από 62 μέλη και μιλώ εξ ονόματος 15 εθνικών αντιπροσωπιών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα αυτή και θεωρούν ότι έχουν ε, πλήρες δικαίωμα να μπορούν ε, να εκφράζονται εντός μιας μεθόδους ε, που θεσπίζει τον κανόνα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή τη μέθοδο DONT. Επίσης, Θέλω να υποστηρίξω αυτή την υποψηφιότητα για διάφορους άλλους λόγους. Καταρχήν, επειδή μιλάμε για ένα πρόσωπο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα του αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ήταν Πρωθυπουργό μάλιστα η κυρία αυτή και μιλάμε και για ε, το ότι έχει ειδικέ αρμοδιότητες ε, σε σχέση με αυτή την Επιτροπή. Επίσης μιλάμε για μια κυρία η οποία ε, ίσως έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους, περίπου μισό εκατομμύριο ψήφους στη χώρα της τις τελευταίες ευρωεκλογές και δεν θα ήταν ε, καθόλου κατανοητόν όλα αυτά τα στοιχεία και οι αιτιολογίε δεν αρκούσαν για την υποστήριξη αυτή τη υποψηφιότητα. Ε, ζητώ λοιπόν εξ ε, του ECR και εξ ονόματος όλης της αντιπροσωπείας μας να μπορέσουν να σκεφτούν όλοι και να μπορέσουν να επιτρέψουν ε, την διεξαγωγή ελεύθερων ε, εκλογών ε, προκειμένου να εκλεγεί η συνάδελφος Σίσρου που υποστηρίζουμε εμείς. Then uh, it would be my question to ask. Uh, uh, να ρωτήσουμε λοιπόν τη συνάδελφο αν δέχεται την υποψηφιότητα.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 Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Κύριος Κάσα. Λοιπόν, έτσι όπως έχουν τα κουμπιά, δεν είναι εύκολο τα νέα μέλη να καταλάβουν πώς λειτουργούν. Καλό είναι λοιπόν να το εξηγήσετε. Μπορεί κάποιοι να μπερδευτούν. Ευχαριστώ κύριε Κάσα. Είναι πολύ σημαντικό σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας. Η κυρία Μπίσοπ έχει στήσει το λόγο. Yes. Good evening everybody. On behalf... Καλό απόγευμα σε όλους, εξ ονόματος της ομάδας μου, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα ήθελα να ζητήσω μυστική ψηφοφορία και φυσικά να εξηγήσουμε και την διαδικασία. Ωραία. Επειδή κάποιοι είναι καινούργοι εδώ, θα κάνουμε δοκιμαστικά μια ψηφοφορία, γιατί πράγματι δεν έχουν διαφορετικό χρώμα τα κουβιά. Ελπίζω όλοι να έχετε βάλει την κάρτα σας στο μηχάνημα. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ωραία. Αν... Να εξηγήσω λοιπόν ότι αν πατήσετε το αριστερό κουμπί, είναι θετική ψήφος με πράσινο χρώμα, υπέρ δηλαδή ψηφίζεται έτσι. Ελπίζω έτσι να το βλέπετε και στο μηχάνημα μπροστά σας. Το μεσαίο είναι η αποχή, με λευκό δηλαδή. Και το δεξί κουμπί είναι το κόκκινο. Αρνητική ψήφος όταν ψηφίζετε κατά. Ελπίζω να τα δοκιμάσατε όλα. Δοκιμάστε τα και πάλι πράσινο υπέρ, λευκό αποχή και κόκκινο κατά. Εντάξει, τα βρήκατε, χρειάζεστε βοήθεια. Εάν όχι, φτάνουμε στο τέλος ε, της δοκιμαστικής ψηφοφορίας, θα περάσουμε στην κανονική για την πρόταση εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την εκλογή της κυρίας Μπεάτα Τσίτσλο ως Προέδρο της Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. And now you see that it's blue because it's a secret vote. Είναι μυστική ψηφοφορία λοιπόν. Okay. Sorry, we have, sorry. sorry, have to do the counting. Do, do it again. Do I have to do the whole voting again? Okay, sorry. Α, συγγνώμη. Κάτι δεν πήγε καλά. Θα ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία εκ νέου, λοιπόν. Please vote now. EPP is one in excess. Mr. Από το ΕΛΚ έχει ψηφίσει ένας παραπάνω. Κύριε Κάσα. Και πάλι έχετε ένα παραπάνω. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 19 ψήφοι υπέρ, 34 κατά και 2 αποχές. Ο κύριος Κάζα. Yes, I propose... Θα πρότεινα, Πρόεδρε, να αναβάλουμε και πάλι την συνεδρίαση για να έχουμε χρόνο να βρούμε μία λύση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεβρούμε μία λύση. Υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνέβη. Κάτι τέτοιο εγώ είμαι νέο μέλος. Όμω για μένα η Επιτροπή επασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι μία από τις πιο σημαντικές επιτροπές στο όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν πρέπει να αναστείλουμε την συνεδρίαση για να γίνουν κάποιες ε, συναντήσεις, να το λύσουμε, εντάξει, αλλά θα ήθελα αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος τρέχει. Και το δεύτερο, αντί να παρουσιάζεται μόνο ένα σημείο υποψήφιο ε, και να καταψηφίζουν ε, τα υπόλοιπα κόμματα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατάλογο των υποψηφίων που να μπορούσαμε να του δούμε πριν από τη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πριν από τη συνεδρίαση. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και κλεισμένων των θυρών ε, και δεν είναι καλό για του ψηφοφόρου. Okay. Ε, Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω το ΕΛΚ γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συναντηθούν και οι συντονιστές των ομάδων και να καταθέσουν μία πρόταση, να υπάρχει και χρόνος να σκεφτούν για να εξεύρουν μία καλή λύση. Γιατί νομίζω ότι όλοι στην αίθουσα ενδιαφέρονται γι' αυτό. Παρακαλώ, ε, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε πει και ξαναπεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί και τηρεί δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα όμως απορρίψαμε μία από τις καλύτερες υποψήφιους. Οι δεξιότητες της, οι αρμοδιότητες τις οποίες ε, έχει ήδη διεκπαιρεώσει είναι κάτι που είναι αδιαμφισβήτητο. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος έπρεπε να εκλεγεί. Χρειαζόμαστε βεβαίως αυτή τη στιγμή ένα διάλειμμα για να δούμε τι θα κάνουμε, μία διακοπή, αλλά πραγματικά απορρίψαμε μόλις μία υποψήφια η οποία πήρε πάνω από 500.000 ψήφους. Τι πιο δυνατή υποψήφιο μπορούσαμε να έχουμε. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ σε αυτή την αίθουσα με αυτή την απόφαση απόρριψης. Διότι αν τηρήσουμε την αρχή της αναλογικότητας, πραγματικά κάτι πρέπει και εμείς εδώ να εκφράσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτή τη διακοπή. Η κυρία Μπίσοπ. Ευχαριστώ. Εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία του κυρίου Κάσα για την διακοπή αυτής της συνεδρίασης. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και εμείς στην πολιτική μας ομάδα βεβαίως και σεβόμαστε όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ομάδα του ECR, αλλά θεωρούμε ότι οι αξίες μας ε, είναι διαπραγμάτευτες και πιστεύουμε ότι οι αξίες είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να στηρίζουν μια αποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την διακοπή και την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Εμείς οι πράσινοι επίσης ζητούμε αυτή την αναβολή. Πρέπει να βρούμε μία λύση από κοινού. Σας ευχαριστώ, κύριε Και το άρθρο 213 του κανονισμού προβλέπει ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και στις επιτροπές αλλά και σε όλα τα όργανα. Αυτό δεν είναι κάτι το προαιρετικό, είναι κάτι το υποχρεωτικό δεσμευτικό και πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά και εδώ και σε αυτή την Επιτροπή να αντικατοπτρίζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η κυρία Ήρτο ζήτησε τον, το λόγο. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να σας ε, ευχαριστήσω που μου δείξατε τέτοια εμπιστοσύνη. Εγώ θέλησα να πάρω το λόγο γιατί ένα μέλος της Επιτροπής μόλις είπε ότι θέλετε κάποιον που να σέβεται τις αξίες, κάποιον που δίνει μεγάλη σημασία στις αξίες. Αυτό που πραγματικά άκουσα με στενοχώρησε, με λύπησε και νομίζω ότι αυτός που πήρε το λόγο και εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο δεν με γνωρίζει. Πραγματικά ανήκω σε... στην ομάδα αυτή των ανθρώπων και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σπάνιο στην αίθουσα που θεωρούν πραγματικά τις αξίες κάτι το θεμελιακό και μέχρι τώρα στην ε, εργασία μου αλλά και σαν Πρωθυπουργό της χώρας μου της Πολωνίας κάθε φορά προσπάθησα είτε σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να εκπροσωπήσω την χώρα μου όπως παραδείγματος χάρη συζητήσεις που χώρα στην ε, Ολομέλεια, πάντα, πάντα στηρίζομαι και κατευθύνομαι από τις ευρωπαϊκές αξίες και θεωρώ πραγματικά κάτι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονό ότι δεν τις ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη εδώ. Και ε, αυτή τη στιγμή δεν μιλώ εξ μου, μιλώ εξ ονόματος όλων αυτών των πολιτών της χώρας μου των 500.000 ψηφοφόρων που με υποστήριξαν, που ψήφισαν για μένα στις ε, ευρωπαϊκές εκλογές. Και όλοι αυτοί στηρίζουν τις προσπάθειές μου, την ε, δουλειά μου στην κυβέρνηση και όλοι ξέρουν ότι πραγματικά εργάστηκα προς όφελος των πολιτών της χώρας μου. Και νομίζω ότι αν αναρωτηθείτε γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη περνάει αυτή την τρομερή κρίση, θα καταλάβετε ότι αν κοιτάξετε τι κάναμε εμείς στην Πολωνία, θα καταλάβετε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παίρνουμε θέσεις που διχάζουν. Και θα πρέπει και για αυτήν εδώ την ψηφοφορία να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί υπάρχει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος έχει δεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι εξ ονόματος της ΚΟΕ εμείς υποστηρίζουμε την αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου να βρούμε έναν υποψήφιο που να μπορέσει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στην Επιτροπή βάσει και του συστήματος DONT. Μάλιστα. Άκουσα λοιπόν ε, πολλές φωνές ε, να ζητούν ε, την διακοπή της συνεδρίασης και την αναβολή της. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε με ένα χειρός. Σας ευχαριστώ που ήλθατε στη συνεδρίαση αυτή. Θέλετε να ψηφίσουμε. Θέλουμε μυστική ψηφοφορία ή όχι. Όχι. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής της συνεδρίασης. Ηλεκτρονικά. Η γραμματεία θα ήθελε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ, λοιπόν, όποιο είναι υπέρ, να πατήσει το πράσινο κουμπί, όποιο είναι κατά. Πράσινο υπέρ της αναβολής και το κόκκινο να το πατήσετε αν θέλετε να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Δεν ψηφίσατε ακόμη όλοι. The, motion is to postpone the meeting and that's in... Λοιπόν, η πρόταση είναι να αναβληθεί η συνεδρίαση. Υπέρ το πράσινο, κατά το κόκκινο. Ψηφίσατε όλοι. Vote is closed. Λήξη. 45 υπέρ της αναβολής της συνεδρίασης. 8 κατά. Σας ευχαριστώ. Και θα σας ενημερώσουμε για τις νέες δυνατότητες ψηφορίας. Ευχαριστώ.